Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Έχετε τα πρακτικά της θεσινή συνεδρίασης ε, στην διάθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί. Περνούμε στο πρώτο σημείο μα. κοινή συζήτηση.